Σουλή και Λουνατσέκ το Κοινοβούλιο ενημερώθηκε ότι από τις 9 Νοεμβρίου 2017 θα χειρεύει θέση τη και με βάση τον κανονισμό ε, ενημέρωσε τις αρμόδιες εθνικές αρχές. Επίσης, η κυρία Λούνατσεκ παραιτήθηκε ε, και από αντιπρόεδρος από τις 24 Οκτωβρίου 2017. Την ε, ε, Πέμπτη θα εκλέξουμε ένα νέο αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θα αντικαταστήσει την κυρία Λούνατσεκ. Ακριβώς γι' αυτό να σα υπενθυμίσω ότι η παρουσίαση των υποψηφιωτήτων θα γίνει την Τρίτη, 24 Οκτωβρίου του 2017, μέχρι τις 6 ώρα θα πρέπει να πάτε στο γραφείο R00101 για την υποβολή αυτών των υποψηφιότητων στο κτίριο Λουίς και θα πρέπει να αποδεχθεί την υποψηφιότητα αυτή το συγκεκριμένο άτομο. άτομο. Η ψηφοφορία θα γίνει την 5η στις 12 η ώρα. Η Επιτροπή